Παρακαλώ, καθίστε. Η Προεδρία θα κάνει μία ανακοίνωση, οπότε σας παρακαλώ ακούστε με. Όπως γνωρίζετε, σήμερα έχουμε την επέτεια της εκεχηρίας με την οποία έληξαν οι εχθροπραξίες μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και γι' αυτό, για να τιμήσουμε την εκεχηρία με την οποία έληξε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, θα τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των εκατομμυρίων Ευρωπαίων που έχασαν τη ζωή τους κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σας ευχαριστώ. Τα πρακτικά της θεσινής συνεδριάσεως είναι στη διαθεσή σας. Αν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, θεωρούνται εγκεκριμένα. Και τώρα περνάμε στις ψηφοφορίες. Ξεκινάμε με την έκθεση της κυρίας Ματέρα για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής